πρακτικά της ε, χθεσινής συνεδρίασης. Ε, ε, σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες έχω και τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχω, ζητή, έχω λάβει εκ μέρους του Συμβουλίου τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση και έχουμε τρεις μήνες ε, για να ε, υιοθετήσει την ε, θέση του το Κοινοβούλιο και θα αρχίσουμε να συζητάμε στα θέματα των ημερησίων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων